Good afternoon, colleagues, and welcome to... Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω σήμερα το απόγευμα. Να καλωσορίσω ένα φιλοξενούμενο, τον κύριο Ταποκό, από τη γραμματεία της Επιτροπής της Οργάνωσης Αφρικανικής Ενότητας. Θα μιλήσουμε επίσης και για τα ορυκτά και μέταλλα από περιοχές προβληματικές. Λοιπόν, πρώτο θέμα είναι η αποδοχή της μερίσιας διάταξης. Υπάρχει μια πρόταση αλλαγή στο σημείο 10 για το JPA. Ο κύριος Γκέρεντς δεν μπορεί να είναι αύριο το πρωί. Και γι' αυτό ζήτησε στο τέλος του απογεύματος την Τρίτη το απόγευμα, όχι σήμερα και όχι αύριο βέβαια το πρωί. Λοιπόν, μπορείτε να δεχτείτε αυτήν την αλλαγή παρακαλώ. Και οι σκιώδεις να γνωρίζουν ότι το θέμα έχει μετακινηθεί αύριο το απόγευμα. Και όχι αύριο το πρωί για τα και. Στο 2. Έγκριση πρακτικών. 17 Οκτωβρίου είναι σε φάκελό σας, αν έχετε αντιρρήσεις, να τις καταθέσετε πριν το τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Αν δεν κατατεθούν συνεδριάσεις, τότε θα θεωρηθούν δεκτές. Ανακοινώσεις Πρόεδρο, έχω ορισμένες ανακοινώσεις. Η πρώτη, όπως γνωρίζετε, ο Επίτροπος Τηλιανίδης είπε ότι αν διοριστεί η πρώτη του αποστολή θα είναι να πάει στην Δυτική Αφρική για το εμπόλα. Και μάλιστα ορίστηκε και συντονιστής για το εμπόλα, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά για το σύνολο της Ένωσης. Θα πάει στην Αφρική λοιπόν αυτή την εβδομάδα. Ελπίζουμε την επόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα να επανέλθει εδώ και να μας παρουσιάσει τα ευρήματά του. Θα επιστρέψει την Κυριακή, θα αναφερθεί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τη Δευτέρα το πρωί και είπε ότι το απόγευμα είναι στην διάθεσή μας, αλλά δεν έχουμε βρει ακόμα αίθουσα. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να ακούσουμε την ίδια μέρα με το Συμβούλιο για τα ευρήματα του κυρίου Στυλιανίδη στην Γουινέα, τη Σιέρα Λεόνε και την Ιγυρία. Ελπίζω λοιπόν αύριο να επιβεβαιώσουμε την αίθουσα και θα σας ενημερώσουμε. Δεύτερη ανακοίνωση είναι μια άλλη συνεδρίαση στις 24 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. Κοινή συζήτηση ανάμεσα στις Επιτροπές ε, Ανάπτυξης για τα θύματα της σεξουαλικής βίας ε, σε περιοχές όπως το η Κεντρική Αφρική και το Ζαΐρ. Κοινή συνάντηση λοιπόν με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Δικαιωμάτων, συγκεκριμένα του, του ανθρώπου. Θα οργανωθεί και μία ακρόαση για την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ανάπτυξη Κάποιοι από τους συναδέλφους έχουν δημιουργήσει ένα intergroup για το θέμα αυτό στις 6.30 και την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο 5G35 θα υπάρξει μια ανεπίσημη ενημέρωση για την έκθεση του Μιλάνου, τη διεθνή έκθεση του Μιλάνου από τον Φράτς Φίσλερ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΞΠΟ Μιλάνου 2015 θα επισκεφτεί έτσι και αλλιώς ή επισκέφτηκε καλύτερα και τις Επιτροπές Γεωργίας και την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και γράφει μια έκθεση για το Συμβούλιο ο κύριος Φίσλε για το τι θα, για το Συμβούλιο μάλλον της έκθεσης, για τη συνέχεια που θα δοθεί στις αποφάσεις και στα τεκτενόμενα στο Μιλάνο. Και πολλοί συνάδελφοι έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να τον συναντήσουν. Θα σας υπενθυμίσουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την συνάντηση με τον Φραντς Φίσλα. Αυτά για τις ανακοινώσεις. Περνάω τώρα στις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν βλέπω τον κύριο Κρέγκ Μακουέιντ. Παρακαλώ το όνομά σας δεν έχω γραμμένο. Δεν έχουμε ανακοινώσεις εξ ονόματος του Μακουέιντ. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περνάμε στο 5, ώρα ερωτήσεων. Δεν έχουν κατατεθεί ερωτήσεις. Ως εκ τούτου συνεχίζουμε λοιπόν στο 6 που είναι Επιτροπή Παρατήρησης Εκλογών στη Μοζαμβίκη. Έχουμε εδώ την κυρία Σαρτζεντίνη που ήταν η υπεύθυνη για την αποστολή παρατήρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να μας παρουσιάσει τα προκαταρκτικά ευρήματα και μπορεί να μας μιλήσει λίγο γενικότερα όλας για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα προγράμματα παρατήρησης των εκλογών γενικότερα. Πολύ μετριοπαθή σας βρίσκω. Ευχαριστώ Λίντα. Ναι. Παραμένω επικεφαλής Τη αντιπροσωπείας παρατήρησης εκλογών στη Μοζαμβική παρόλο που ήταν στις 15 Οκτωβρίου τρεις εκλογές ταυτόχρονα προεδρικές, βουλευτικές και περιφερειακές, επαρχιακές. Έχουμε μία παράδοση ε, οι ε, αποστολές παρατήρησης εκλογών ευρωπαϊκές να έχουν επικεφαλής έναν ευρωβουλευτή. Τώρα αναλαμβάνει η κυρία Μογκερίνη να διορίζει. Εγώ είχα διοριστεί ακόμα από την κυρία Άστον. Ε, μετά από μια διαβούλευση εδώ στην Επιτροπή που δεν ήταν πάρα πολύ δημόσια, αλλά εσείς συμπροεδρεύσατε ε, μαζί με την Επιτροπή ΑΦΕΤ, νομίζω ονομάζεται ε, Ομάδα Παρατήρησης Δημοκρατικών Εκλογών, κάπως έτσι, εγώ εκεί εκπροσωπώ τους Πρασίνους. Απαρτίζεται από ένα πυρήνα ε, αυτή η Επιτροπή είναι ο επικεφαλής και ο αναπληρωτής που βασικά αναλαμβάνει όλη τη διοργάνωση ε, διότι πηγαίνει στη χώρα, παραμένει εκεί επί και ε, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα πράγματα εκεί μαζί με κάποιον ειδικό εκλογό, λόγο, ας πούμε, ειδικό για τις εκλογές, κάποιον ειδικό για θέματα ενημέρωσης, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη δημοσιότητα των εκλογών συνήθως ε, στον τοπικό τύπο. Ε, και ε, βοηθάει και όλες τις αποστολές και τους νομικούς και την βραχία βραχυπρόθεσμη μάλλον επιτροπή παρατήρησης και τη μακροπρόθεσμη και ε, κανονίζει τα πάντα. Αυτή τη φορά στη Μοζαμβίκη δεν υπήρχε ε, παρουσία ε, αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό έχει να κάνει με τις προτεραιότητες εδώ στο Κοινοβούλιο που είναι η Μολδαβία και η Ουκρανία. Κρίμα. Εγώ προσπάθησα να το αλλάξω αυτό διότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο είχαν συμμετοχή από τις πρώτες εκλογές μετά τον εμφύλιο στη Μοζαμβίκη που έγιναν το 1994 είναι και πολύ διαφορετικός ο τρόπος πλέον ε, που χρηματοδοτείται η ε, ομάδα παρατήρησης των εκλογών. Ε, χρηματοδοτήθηκε από διάφορα κράτη-μέλη της Ένωσης που έχουν πρεσβεία στο Μαπούτο, την πρωτεύουσα της Μοζαβίκης, καθώς το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν λεφτά. Διότι ξέρουμε αυτή την ιστορία με την ανάληψη υποχρεώσεων και τι δαπάνε. Δηλαδή κάπου είχαν δεσμευτεί τα κονδύλια, αλλά για να δαπανηθούν δεν βρέθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, ήταν πολύ σημαντικό έτσι κι αλλιώ να παραμείνουμε, να έχουμε μια παρουσία παρατήρηση ε, εκλογών. Γι' αυτό έβαλαν το χέρι στην τσέπη τα κράτη-μέλη για να πάμε εκεί. Και τελικά είχαμε 20 παρατηρητέ ε, ε, που έμειναν εκεί αρκετό διάστημα και 20 που ήταν βραχυπρόθεσμη η αποστολή ε, που ήταν μια εβδομάδα ε, πριν και μετά τις εκλογές ενώ οι άλλοι ε, μακροπρόθεσμοι ήταν ένα μήνα εκεί. Είχαμε λοιπόν και συνοδοί από διάφορες πρεσβείες και τελικά ήταν πάνω από 100 οι παρατηρητές μας και παρουσία είχαμε σε όλες τις επαρχίες. Τώρα, να σας πω τι έκανα εγώ ως επικεφαλής. Επισκέφτηκα τη χώρα τρεις εβδομάδες πριν από τις εκλογές για να εξοικειωθώ εκεί με την κατάσταση, το Υπουργείο να γνωρίσω τους βασικούς φορείς, το Συνταγματικό Συμβούλιο και την Εφορευτική Επιτροπή, τα διάφορα πολιτικά κόμματα. για να καταλάβουν οι πάντες ότι μας είχαν προσκαλέσει οι αρχές της χώρας, η κυβέρνηση της Μοζαμβίκης. Μόνο έτσι εννοείται ε, επίσημη παρατήρηση εκλογών. Υπάρχουν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές. Λοιπόν, η κυβέρνηση μας είχε ε, προσκαλέσει και ε, πληρούνται όλα τα κριτήρια και τα πρότυπα. Δύο μέρες, στη μεθεπομένη των εκλογών, εξέδωσα μια πρώτη δήλωση προκατακτική Μπορεί κάποιοι να θεώρησαν και να περίμεναν ότι οι εκλογές ήταν ελεύθερες, δίκαιες, αξιόπιστες ή όχι, αλλά έχουμε ξεφύγει εμείς πια από αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Ε, δεν κρίνουμε, δεν αξιολογούμε τις εκλογές. Εγώ είπα ότι ήταν κανονικές ε, οι εκλογές την ίδια την ημέρα, αλλά δεν ήταν ε, ίση, ήταν άνιση η προεκλογική εκστρατεία, γιατί οι εκλογές δεν κρίνονται τη μέρα της κάλπης, αλλά και προεκλογικά. Ε, υπάρχουν διάφορες διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούνται και πάλι κάποια ελάχιστα κριτήρια, αλλά που ίσχυε αυτό, υπήρξαν κάποια επεισόδια και μάλιστα βία σε ορισμένες περιφέρειες αλλά αυτό δεν επηρέασε τις εκλογές στο σύνολό τους, ώστε να χαρακτηριστούν αντικανονικές. Αλλά η προεκλογική εκστρατεία ήταν ετεροβαρής, ε, δεν είχε ισορροπία. Τρία ήταν τα κόμματα με τρεις υποψηφίους για το αξίωμα του Προέδρου. Φρολίμο, η κυβέρνηση, Ρενάμο, η αξιωματική αντιπολίτευση και ένα κόμμα που παίζει ήδη ρόλο και έπαιξε ε, ε, στο παρελθόν, στον φίλιο ε, πόλεμο και ένα νέο κόμμα, MDM, που είναι ένα κόμμα που έχει αποσπαστεί από ένα από τα προηγούμενα και προσελκύει ψηφοφόρους νεότερους και από αστικές περιοχές κυρίως. Το κόμμα Φραλίμο χρησιμοποιούσε τις κρατικές υποδομές και το Ρενάμο τοπικό επίπεδο, αλλά κυρίως το Φραλίμο. Ε, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ήταν δίκαιη η κατανομή, πώς να το πω, των δυνατοτήτων. Είχαν λοιπόν συγκριτικό πλεονέκτημα και άδικο τα μέλη του ενός κόμματος σε σχέση με τα άλλα δύο. και κάναμε και μια έρευνα για τα βασικά μέσα ενημέρωσης, κρατικά, ιδιωτικά, ανεξάρτητα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπο. Ε, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης βεβαίως ήταν ε, ε, μεροληπτικά υπέρ του κυβερνώντος κόμματος. Μετά από όλα αυτά όμως δεν τελείωσαν οι εκλογές. Εγώ έφυγα λίγες μέρες αργότερα. Η μακροπρόθεσμη αποστολή παρέμεινε και ο πυρήνας που έμεινε μέχρι την περασμένη Τετάρτη και την Πέμπτη του συνάντησα στις Βρυξέλλες για την ενημέρωση στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Αλλά μετά την καταμέτρηση των ψήφων στην εκλογική νύχτα, που ήταν επίσης αρκετά ε, κανονική, θα έπρεπε να γίνει μια αναγωγή και να συγκεντρωθούν τα αποτελέσματα και αυτό πήρε πάρα πολύ χρόνο. Προσπάθησαν οι δικοί μας παρατηρητές να έχουν πρόσβαση ε, στα κέντρα που είχαν ε, συγκεντρώσει τα αποτελέσματα. Αυτό έγινε αποσπασματικά όμως και μόλις πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα αν δεν απατώμε, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μας έδωσε το επίσημο αποτέλεσμα των εκλογών που συμφωνούσε με την εναλλακτική καταμέτρηση που έκανε η κοινωνία των πολιτών και κέρδισε τις εκλογές ο, ο πρόσωπος του Φραλίμου, ο υποψήφιος, 57% νομίζω πήρε και το Ρενάμο και το MDM, τα άλλα δύο κόμματα απογοητεύτηκαν από το αποτέλεσμα και υπήρξαν και πολλές καταγγελίες στη συνέχεια. Ε, και ενστάσεις. Δεν έχουμε όμως τελικά το οριστικό αποτέλεσμα, διότι έγιναν αυτές οι ενστάσεις προς και οι προσφυγές του Συνταγματικό Δικαστήριο και από τα δύο κόμματα, και το Ρενάμο και το MDM. Νομίζω μάλιστα το Ρενάμο ζητάει ακύρωση κανονικά των εκλογών σε κάποιες επαρχίες, το ίδιο και το κόμμα MDM, και μόνο εφόσον αποφανθεί το Συνταγματικό Συμβούλιο, που θα ανακοινωθούν τα επίσημα αποτελέσματα και από τότε μόνο και πέρα θα βγάλω εγώ την τελική μου έκθεση. Γιατί το κάνουμε αυτό. Γιατί θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι λαμβάνουμε υπόψη όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Προεκλογικά, την ημέρα των εκλογών και μετεκλογικά. Διότι αυτές οι εκλογές έχασαν την αξιοπιστία και το κύρος τους μόνο αφού του έγιναν. Αυτό βεβαίως είναι μια απογοήτευση, αλλά μπορεί κανείς ε, να το εξασφαλίζει μόνο παραμένοντας ε, επί τόπου, ε, γιατί δεν έχει τελειώσει η κατάσταση πριν ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, για πρώτη φορά εγώ να αναλάμβανα αυτά τα καθήκοντα, μελέτησα πάρα πολύ το σύστημα Βλέπετε τις ομοιότητες και τις διαφορές πάντα σε σχέση με τα όσα κανείς ε, γνωρίζει. Και κάτι που ήταν ενδιαφέρον πλην ανησυχητικό. Το εκλογικό σύστημα, ο εκλογικός νόμος δηλαδή στη Μοζαμβική είναι άκρος πολιτικοποιημένος σε όλα τα επίπεδα και στο Συνταγματικό Συμβούλιο και στην Εφορευτική Επιτροπή ε, ακόμα και στα ίδια τα εκλογικά τμήματα είχαμε εκπροσώπους παρόντες των τριών πολιτικών κομμάτων και με ρόλο μάλιστα. Είχαν πει όλα τα κόμματα ε, και μάλλον έτσι νόμιζαν ότι εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά την ίδια τη μέρα των εκλογών είναι δύσκολο ε, αυτά να εφαρμοστούν, γιατί είναι 17.000 τα εκλογικά τμήματα. Και να έχεις παντού μέλος ε, και στην Επιτροπή εκεί του, του εκλογικού τμήματος και εκπρόσωπο κομματικό, εκλογικό. Για τα δύο μικρά κόμματα ήταν πολύ μεγάλη αυτή η επιβάρηση να έχουν 17.000 εκπροσώπους. Και μετά έπρεπε να συναντηθούν και να συμφωνήσουν ότι αυτή είναι η διαδικασία. Τελικά παρέλυσε αυτή η διαδικασία και διχάστηκε και η Φορευτική Επιτροπή, η Κεντρική, ε, ανάλογα με το σε ποιο κόμμα ανήκει κάθε μέλος. Τώρα πρέπει να δουν πώς θα συνεχιστεί αυτό το πολιτικοποιημένο σύστημα. Μπορεί να προχωρήσει η χώρα βέβαια σε κάποια πολιτικοποίηση, αλλά δεν θα είναι τόσο ανεξάρτητη, γιατί το κόμμα ταυτίζεται με το κράτος και τούμπαλι. Αλλά και πάλι εγώ παρατηρήτρια είμαι και τίποτα άλλο, δεν συμμετέχω εκεί σε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ, Τζούντιθ, για την πληρέστατη παρουσίαση και της διαδικασίας και του τι έγινε στη Μοζαμβίκη. Καταλαβαίνω το δίλημα στο τέλος. Πραγματικά είναι δύσκολο για τα πολιτικά κόμματα, ακόμη και στις δικές μας ε, χώρες που μπορεί να είναι σε όλα τα εκλογικά τμήματα. Είναι τεράστιο το ε, εγχείρημα. Και υπάρχουν και κάποιες χώρες που δεν το επιτρέπει η το επιτρέπει, τέλο πάντων είναι δύσκολο. Γκερέρο Σαλόμ. Δεν θέλω να κάνω ερώτηση. Να συγχαρώ θέλω την κυρία Σαρτζεντίνη πρώτα απ' όλα για τις εξηγήσεις που μας έδωσε σε σχέση με την εκλογική διαδικασία στη Μοζαμβίκη, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια εκλογική διαδικασία με τέτοια χαρακτηριστικά. Η κυρία Σαρτζεντίνη έκανε και την αξιολόγησή της, παρουσίασε την κατάσταση ως προς το τι έγινε πριν τις εκλογές, τι έγινε την ημέρα των εκλογών και ως προς το κατά όσο μπορεί να γίνει αποδεκτό από τους πολίτες ε, συνολικά, το σύνολο μάλλον της εκλογικής διαδικασίας αυτής. Είδα την ανακοίνωση τύπου, δεν ξέρω τώρα αν έκανα λάθος, νομίζω 6 Νοεμβρίου. Ήταν 15 ε, Οκτωβρίου έγιναν οι εκλογές. Άρα υπήρξε ένας χρόνος ορίμανσης. Δεν αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα το εκλογικό την επομένη ακριβώς ή το βράδυ των εκλογών. Γιατί πολλοί ήταν έτοιμοι ίσως να επιστρέψουν στις χώρες τους ή στις Βρυξέλλες εκείνο το βράδυ. Πέμπτες στη σειρά οι εκλογές αυτές στη Μοζαμβίκη όταν και αφού το έληξε ο εμφύλιος πόλεμος. Άρα έχουμε μια κάποια σταθερότητα πια συγκριτικά με το πώς έχει κατάσταση σε πολλές άλλες ε, περιοχές της Αφρικής. Αυτό σημαίνει κυρίως ότι πρόκειται για μια σταθερότητα πάντοτε βέβαια πρέπει να και να διατηρηθεί και να βελτιωθεί. Το κράτος πρέπει να είναι ανοιχτό, και να υπηρετεί τους πολίτες. Θα ήθελα να κάνω κανένα δύο σχόλια τώρα για τις επιτροπές ε, παρατήρησης εκλογών. Ναι, μεν μας έχουν προσκαλέσει, ουσιαστικά, μάλλον μας έχετε εσείς ζητήσει ουσιαστικά να το κάνουμε. Εγώ έχω συμμετάσχει σε τρεις τέτοιες επιτροπές παρατήρησης εκλογών. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες αντιπαραθέσεις και προβλήματα. Από τις τρεις Μόνο στην Κένια ήταν κάπως πιο χτυπητό το πρόβλημα, ας πούμε. Όπως είπε και η Τζούντιθ. Έτσι και στην περίπτωση αυτή δεν υπήρχε αποστολή του Κοινοβουλίου, αλλά της Ένωσης. Συνήθως όμως υπάρχει η Επιτροπή του Κοινοβουλίου, η οποία είναι ένα κομμάτι της αντιπροσωπείας της Ένωσης και οι προσωπίες αυτές είναι, χαρακτηρίζονται από μεγάλο επαγγελματισμό. Δηλαδή όσοι παραμένουν ε, για μακρόχρονικό διάστημα, οι λεγόμενοι μακροπρόθεσμοι, μακροχρόνοι παρατηρητές μπορούν να δώσουν πολύτιμη περιγραφή για το τι συνέβη, ποια είναι η νομική συνταγματική εκλογική δομή της χώρας, και να κάνουν μια πολύτιμη αξιολόγηση. Όπως είπε η Τζούντιθ, τα μεγαλύτερα προβλήματα συνήθως ε, προκύπτουν πριν την ημέρα των εκλογών, έχουν να κάνουν ε, με την ε, απογραφή. Κάποιες φορές υπάρχουν προβλήματα γιατί πολλές φορές στους εκλογικούς καταλόγους εγγράφονται περισσότεροι από αυτοί που έχουν δικαίωμα και οι κάρτες εκλογικές μπορεί να αργήσουν να φτάσουν στους δικαιούχους ε, και έτσι δημιουργούνται ακόμη περισσότερες δυσκολίες. Η κατάσταση σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα μέσα επικοινωνίας μπορεί να είναι ασύμετρη, να μην είναι ισοδίκαιη και με τα προβλήματα αυτά βέβαια δημιουργείται ανισότητα, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι, στην εκλογική αναμέτρηση. Για να σας ε, μεταδώσω ουσιαστικά τη δική μου εμπειρία. Σε αυτές τις επιτροπές παρατήρησης εκλογών διατρέχουμε ένα κίνδυνο να είμαστε υπερβολικά απαιτητικοί στη χώρα που γίνονται εκλογές για κάποια θέματα που στις δικές μας χώρες μπορεί να μην είναι τόσο επεκτικά. Δηλαδή, εάν συζητήσουμε στις χώρες μας συζητήματα που έχουν να κάνουν με την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων, που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης για τους διάφορους υποψηφίου. αν συζητήσουμε τη διαφορετική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων κτλ. κτλ. Ε, το να μπορούμε να κάνουμε μαθήματα σε άλλες ε, χώρες ε, νομίζω θα καταλαβαίναμε ότι δεν είναι και πάρα πολύ σκόπιμο. Θέλουμε να τηρούνται τα δημοκρατικά κριτήρια, τα βασικά δημοκρατικά κριτήρια, δηλαδή να αγωνίζονται ισότιμα όλοι οι συμμετέχοντες στις εκλογές, αλλά καλό είναι πρώτα να βλέπουμε τα του οίκου μας, τι γίνεται στις δικές μας χώρες και αν είναι τόσο τέλεια κατάσταση σε εμάς. Είμαι Ισπανός, Έχω λάβει μέρος και σε κάποιες άλλες, έχω παρατηρήσει μάλλον εκλογές όπως το Πέρου για παράδειγμα. Είχαμε κάποιες επιφυλάξεις για το άνοιγμα των εκλογικών τμήματων, την ε, ε, διανομή των ψηφοδελτίων. Ήταν επιφυλάξεις θεμητές και δικαιολογημένες. Κατά πάσα πιθανότητα όμως ε, σε πολλά ισπανικά χωριά τη μέρα των εκλογών θα μπορούσε κάποιος να αναφέρει ακριβώς τις ίδιες επιφυλάξεις. Υπάρχει και το εξή θέμα, ότι εκ των προτέρων ε, θεωρούμε αξιόπιστα τα δικά μας εκλογικά συστήματα και εκ των προτέρων θέτουμε επιφυλάξεις για άλλα συστήματα που ή λειτουργήσαν κακά ε, ε, λάθος στο παρελθόν ή το επίπεδο δημοκρατικής εδραίωσης, παγίωσης είναι μικρότερο στις περιπτώσεις αυτές από τις δικές μας χώρες. Από αυτήν την έννοια οι παρατηρήσεις και η δήλωση τύπου, γιατί περιμένουμε ακόμη την οριστή έκθεση της κυρίας Νομίζω είναι κατάλληλα, ε, κατάλληλες οι ενδεδειγμένες αυτές οι διατυπώσεις. Ξέρουμε ότι υπάρχει κώδικας δεοντολογίας για τα μέλη των Επιτροπών Εκλογικής Παρατήρησης. Και βέβαια το βασικό εκεί είναι η ουδετερότητα, η αμεροληψία. Πολλές φορές τίθεται ε, να αυτή η ουδετερότητα και από την ίδια την κοινοβουλευτική ιδιότητα. Δεν θα σας πω ε, κάτι καινούργιο, αν σας πω ότι υπάρχουν κάποιοι οποίοι καίγονται να κάνουν δηλώσεις στο CNN και στο BBC τη μέρα των εκλογών για να δουν αν θα βγουν ε, στο γυαλί ε, στη χώρα τους. Άλλοι τηρούν βέβαια τα τα δέοντα ανάλογα με τον κοινοβουλευτικό ρόλο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε υποδειγματικοί, τουλάχιστον σε τέτοιες περιπτώσεις, στις χώρες που πηγαίνουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ Νρίκη. Πρέπει να σας πω για τη χώρα μου ότι εμείς δεν έχουμε κάποια είδος ταυτότητας ή κάρτας ε, για να ψηφίσουμε, απλά παρουσιαζόμαστε στο εκλογικό τμήμα και ψηφίζουμε. Αυτό φαντάζομαι ότι το βρείτε περίεργο εσείς, αλλά ε, μόνο σε ένα τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου έχει δημιουργήσει αυτό πρόβλημα. Ε, τώρα το να φάμε ε, ε κάποιοι, για σας μπορεί να ήταν πολύ περίεργο και να φόβησε και κάποιος το να πάνε κάπου να ψηφίσουν χωρίς να έχουν ένα τρόπο ταυτοποίησης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μια που μιλάμε για διαφορετικές κουλτούρες και παραδόσεις και ιδιοσυγκρασίες, έλεγα, Πρόεδρε, μια που μιλάμε για αυτά τα θέματα, ιδιοσυγκρασίες λαών, παραδόσεις και κουλτούρες, να σας πω κάτι μιλώντας πορτογαλικά. Μας ενώνει η ίδια γλώσσα με τη Μοζαμβίκη. Θέλω να πω ότι είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες προς την κυρία Σαρχεντίνη για τη δουλειά της και ε, γενικά ε, σε όλη την Επιτροπή Παρατήρησης ε, Εκλογών αξίζουν συγχαρητήρια και ευχαριστίες. Η έκθεση της είναι προσωρινή, όπως είπε και η ίδια. Δεν είναι η οριστική. Ξέρουμε ότι ήταν πολύ μεγάλη αντιπαράθεση στις εκλογές, γιατί υπήρχαν και διαμαρτυρίες και κατηγορίες που κατέθεσαν και ενστάσεις τα πολιτικά κόμματα σε σχέση με τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας κάνει να λησμονούμε τις προόδους που έχει επιτελέσει η χώρα στον εκδημοκρατισμό και στην ε, εκλογική διαδικασία. Το τονίζει αυτό η έκθεση, ότι επιτέλους ε, υπάρχει ε, μία συμφωνία για την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων με βάση την απογραφή που στηρίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, Μπορεί να ήταν άνηση και μεροληπτική η προεκλογική εκστρατεία, ήταν ε, όμως ειρηνική. Και την ίδια την ημέρα των εκλογών πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ειρηνική εκλογική ημέρα χωρίς μείζωνα επεισόδια. Επίσης θέλω να πω εδώ ότι μέσω αυτών των εκλογών ε, αναδύθηκε ένα νέο πολιτικό κόμμα με σημαντική απήχηση στο εκλογικό σώμα. Αυτό λέει πολλά για το υψηλό δημοκρατικό φρόνημα και επίπεδο γιατί γνωρίζετε ότι οι χώρες σε μεταπολεμικές ή μετεμφυλιακές ε, καταστάσεις ε, γνωρίζουν τέτοια προβλήματα και πολλά ακριβώς λόγω των εμφυλίων. Το γεγονός λοιπόν ότι τώρα αναδύονται νέα κόμματα και ήρθαν και ψήφισαν πολύ αυτό το νέο κόμμα, ε, είναι ενθαρρυντικό και θετικό. Γιατί είναι νεαρή η δημοκρατία στη Μοζαμβίκη ακόμα. Εν πάση περιπτώσει αμφισβητήθηκαν τα αποτελέσματα, θα πρέπει να διασκεδαστούν αυτές οι αμφιβολίες και οι ανησυχίες. Πάντως η δική μας αντιπροσωπεία πολύ καλά κάνει να μην εκδίδει την τελική ε, έκθεση, διότι εκκρεμούν ακόμα εκεί τα πράγματα και οι καταστάσεις. Λοιπόν, θα πρέπει να περιμένουμε να πάρει το δρόμο της η διαδικασία αυτή. Α, γνωρίζετε κατά τα άλλα ότι είναι και αυτό το τμήμα της εκλογικής διαδικασίας, η αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων των εκλογών. Και γι' αυτό θα πρέπει να εξεταστεί πρώτα η κάθε έσταση και μετά να βγάλει το πόρισμα ή την έκθεσή της η Επιτροπή μας. Αυτό είναι και ένα τμήμα, αν θέλετε, μιας ε, εκλογικής διαπαιδαγώγησης και ενίσχυση του κράτους δικαίου και γενικότερα των πολιτικών ε, και ε, αστικών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Κύριος Νόησερ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά καταρχάς και εγώ την κυρία Σαρχεντίνη, κυρίως γιατί πήγε και νωρίτερα ε, και ε, δραστηριοποιήθηκε και εκτός της Επιτροπής. Όποιος τη γνωρίζει την κοινότητα της Αρχεντίνη ξέρει πόσο ε, εντατικά προετοιμάζεται και με ποια επιμέλεια. Ζήτησα όμως το λόγο διότι έχω προβλήματα με τη διαφορά με την οποία αντιμετωπίζουμε την παρατήρηση εκλογών. Εγώ ήμουν παρατηρητής στην Ουκρανία και όταν έκλεισαν οι κάλπες και τα εκλογικά τμήματα τη Δευτέρα το πρωί ήδη έπρεπε να δώσουμε τη γνωμοδότησή μας. Και μου άρεσε πολύ αυτό που είπε η Γιούντιτ, ότι βγάλαμε μια γνωμοδότηση με την ησυχία μας να καταραγιάσει λίγο ε, η φασαρία, να συλλέξουμε στοιχεία θέλαμε και μετά να βγάλουμε. Στην Ουκρανία τελείω διαφορετική η γνώμονε και τα κριτήρια. Και καλά θα κάναμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά παντού σε όλε τι αποστολέ παρατήρηση εκλογών. Τουλάχιστον θέλω να το πω να σημειωθεί αυτό. Τώρα, έρχομαι στο δεύτερο σκέλος της τοποθέτησής μου που είναι ερώτηση. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε καλή συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση και τις χώρες ΑΚΕ. Και ξανά και ξανά αναδύεται και η ιδέα που εν μέρει έχει εφαρμοστεί κιόλα να κάνουμε κοινέ παρατηρήσεις εκλογών με την Αφρικανική Ένωση, με τις χώρες Αφρικής, Καραβικής, Ειρηνικού. Και έρχομαι τώρα να ρωτήσω. Καλά, αυτή ήταν τώρα μονομένη ε, παρατήρηση εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε επαφές με παρατηρητές της Αφρικανικής Ένωσης ή των χωρών ΑΚΕ. Γιατί καλό θα ήταν και σε αυτό το επίπεδο να προσπαθήσουμε να συντονιστούμε και να συγκλίνουν κάπως τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε και τα μέτρα και τα σταθμά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η υπηρεσία εξωτερική δράση Είναι εδώ κανεί παρόν και θέλει να πει τίποτα. Παρακαλώ. Και μετά η κυρία Σαρχεντίνη. Ευχαριστώ Πάολο Σάλβια από το Τμήμα Παρατήρηση τη Δημοκρατία Εκλογών τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, απαντώντα στο τελευταίο σημείο για τη συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση, ορίστε δίπλα μου το σαφέ παράδειγμα μιας εταιρική σχέσης και συνεργασίας ε, με τις ε, χώρες αυτές, αλλά και με άλλε περιφερειακές οργανώσεις. Ε, πρέπει να σα πω ότι πράγματι κοινή δουλειά γίνεται, είναι κανονική πλέον διαδικασία και πρακτική να υπάρχει μια μόνιμη ανταλλαγή πληροφοριών και μόνιμη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών αντιπροσωπιών, Αφρικανική Ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε μικτές επιτροπές παρατήρησης, αλλά είναι κάτι που το σκεφτόμαστε σε ορισμένε περιπτώσεις και στο μέλλον θα μπορούσε να είναι μια δυνατότητα, τουλάχιστον προς διερεύνηση. Πέραν όμως αυτής της ιδέας ε, να έχουμε μια κοινή μεικτή αντιπροσωπεία, έχουμε συνεργασία η οποία δεν αφορά μόνο ε, την επιτόπου συνεργασία που έχουμε στις εκλογές, και με την ΕΚΟΒΑΣ και με την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης έχουμε πολύ καλή συνεργασία και μάλιστα προβήκαμε και σε κοινέ δηλώσεις μία μέρα πριν από τις εκλογές καλώντας ε, όλους τους μετέχοντες να σεβαστούν τις διαδικασίες αλλά υπάρχει και ε, συνεργασία, θα το επαληθεύσει ο συνάδελφος ε, και γενικότερα δηλαδή έχουμε την κατάρτιση, την εκπαίδευση των παρατηρητών των εκλογών. Είναι ένα πρόγραμμα που το εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα πολλοί από τους παρατηρητές ε, επιτόπου έχουν εκπαιδευτεί ε, στο πλαίσιο αυτού του, του κύκλου μαθημάτων. Σίγουρα η συνεργασία μας έχει βελτιωθεί τα μάλα σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Τζούντιθ. Ε, ε, uh, Δύο σχόλια και μία απάντηση στον κύριο Νόισερ. Νομίζω ο κύριος Γκερέρο είπε κάτι για την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Ε, διαπίστωσα με ενδιαφέρον ότι 90% ε, είναι η συμμετοχή, δηλαδή πηγαίνουν οι πολίτες και δηλώνονται για να εγγραφούν σε εκλογικό κατάλογο. Αλλά υπάρχει λόγος γι' αυτό. Είναι πολύ πιο εύκολο να πάρεις ε, εκλογικό βιβλιάριο, ας πούμε, κάρτα εκλογέα, παρά ε, αστυνομική ταυτότητα. Και έχεις λοιπόν αυτή την κάρτα εκλογέα και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις ως ταυτότητα. Ε, ε, αλλά η εγγραφή ήταν υψηλή, η συμμετοχή ήταν χαμηλή, 50%. Απογοητευτικό αυτό. Μετά τις εκλογές τώρα στη Μοζαμβίκη, τι διαπιστώνουμε. Ο νέος πρόεδρος δεν έχει ισχυρή νομιμοποίηση. Μάλλον όχι. Δεν είχε προσωπική συμμετοχή στον εμφύλιο πόλεμο, ούτε συνδέεται ε, με αυτό. Για πρώτη φορά και για όλη την Νότια ε, ε, το νότιο τμήμα της Αφρικής. Έχει σημασία αυτό. Σκεφτείτε το Ζούμα στη Νότια Αφρική και τον ε, Μουγκάμπε στη Ζιμπάμπουε ε, και την Αμιμπία. Δηλαδή είναι ένας ε, πρόεδρος τώρα ετών γύρω στα 50 που δεν έχει συμμετάσχει στον εμφύλιο πόλεμο ότι μπορεί κανείς να του προσάψει κάποια συμμετοχή. Δεν ξέρω ποια είναι τα πολιτικά του σχέδια διότι μετά από αυτή την προσεκτική παρατήρηση των εκλογών ακόμα δεν έχω καταλάβει τα πολιτικά σχέδια των τριών μεγάλων κομμάτων. Δηλαδή τι, τι ενθάρρυνε, τι κινητοποιούσε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει τον έναν ή τον άλλον. Ε, για τη συνεργασία Νόρμπερτ, εγώ ε, συνάντησα τους επικεφαλείς της ΣΑΝΤΕΚ, ε, της Αφρικανικής Ένωσης, ΆΙΣΑ και ε, τις ε, πορτογαλόφωνες χώρες και άλλους. Ε, για μένα σημασία έχει η αποστολή μας να συνεχίσει να δραστηριοποιείται με έναν τρόπο πάρα πολύ ανεξάρτητο. Διότι οι συνάδελφοι των άλλων επιτροπών παρατήρησης πολύ γρήγορα, δύο μέρες μετά έλεγαν ότι ήταν όλα εντάξει, μια χαρά πήγαν οι εκλογές. Εγώ την επομένη των εκλογών το πρωί συναντήθηκα με όλους τους επικεφαλείς, με, με επικεφαλής έναν υπουργό της Νοτιού Αφρικής που εκπροσωπούσε τη ΣΑΝΤΕΚ και είχα την αίσθηση ότι να βγάλουμε ε, ανακοίνωση ήταν, ότι ήταν ωραία όλα και πεντακάθαρα. Ήταν πολιτικό ε, πολιτικός υποκινούμενη δήλωση. Και εγώ θέλω, ήθελα να συνεργαστούμε όσο γίνεται περισσότερο, να προσπαθήσουμε να έχουμε δηλώσεις ε, συντονισμένες, ενωμένες, αλλά χωρίς πολιτικά κίνητρα. Okay, thanks very much. Um, Ευχαριστώ πολύ την Τζούντιθ Σαρτζεντίνη και για την έκθεση και γιατί ήρθατε εδώ σήμερα. Ε, Τζούντιθ, περνάμε στο σημείο 7 μιλάμε για μεταλλεύματα που προέρχονται από περιοχέ συγκρούσεων. Θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων, αφού ακούσουμε όμω πρώτα τον κύριο Βέντα, τον συντάκτη Γνωμοδότηση από την Επιτροπή μα. Να σα ενημερώσω σχετικά, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η Επιτροπή μα και οι συντονιστέ συγκεκριμένα θεώρησαν ότι το ζήτημα αυτό των μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχέ συγκρούσεων έχει ε, μια σημαντική ε, πτυχή ε, και περιβαλλοντική. Εμείς ζητήσαμε να είμαστε υπεύθυνοι ε, για τα περί του άρθρου 55, η τα είναι η αρμόδια καθήλυνη. Θέλαμε να έχουμε πλήρη συναρμοδιότητα. Μετά αναφέραμε το άρθρο 54, όσο μου κυβάσει πάω ούτε αυτό ε, δεν το δέχτηκαν για να είμαστε συνδεδεμένη επιτροπή. Στην επιτροπή τα δεν το έχουν δεχθεί ακόμη. Και με την Επιτροπή Εμπορίου δεν έχουμε ακόμη καταλήξει. Άρα αυτή τη στιγμή προχωράμε με μια κανονική γνωμοδότηση, την οποία καταρτίζει ο κύριος Βέντα. Έγινε μια αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα. Θα σας το πω στη... στο τέλος. Γιατί δίνει έναν παραπάνω μήνα ίντα τώρα. Θα σας πω όμως πως έχει το χρονοδιάγραμμα. Είναι μεγάλη περίοδος που έχουμε μπροστά μας. Βέβαια, οι πρόεδροι των ε, επιτροπών στη διάσκεψή τους θα τα αποφασίσουν. Η Τζούντιθ έχει ζητήσει ω σκιώδη ε, των ε, Πρασίνων και επειδή πρέπει να πάει στι 5 σε ένα τριμερή διάλογο, έχει ζητήσει το λόγο. Αν λοιπόν ε, δεν έχετε αντίρρηση, να προηγηθεί κυρία Σαρτζεντίνη των άλλων εισηγητών και σκιωδών. Ο κύριος Βέντα ως εισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω την τιμή να είμαι εισηγητής για αυτό το θέμα, το οποίο έχετε και σας απασχολήσει και σας σχετικά με την εισαγωγή των ορυκτών τανταλίου, βολφραμίου και όπως είπε η κυρία Μακάβαν, η πρόεδρός μας, συνδέονται διάφορα τεχνικά θέματα με τις αρμοδιότητες της κυρίας Επιτροπής επί της ουσίας. Εμείς θα πάρουμε την τελική απόφαση, την απόφαση επί της ουσίας για τον μελλοντικό κανονισμό. Συνεργαστήκαμε λοιπόν με την Επιτροπή Ίντα, είχαμε μια καλή συνεργασία, με προσκάλεσαν και σε μια συνεδρίασή τους και αυτός ο κανονισμός έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την Επιτροπή Ανάπτυξης. Dla chciałem powiedzieć, że w dniach 3 i 4 grudnia w Komisji INTA ma się odbyć Στις 4 λοιπόν Δεκεμβρίου θα οργανωθεί στην ΙΝΤΑ και μια δημόσια ακρόαση για το συγκεκριμένο αυτό θέμα των ορυκτών προϊόντων στις ζώνες συγκρούσεων ε, το θέμα είναι η σχέση που έχει η επεξεργασία και η εκμετάλλευση κυρίως αυτών των ορυκτών με ε, τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στις περιοχές εξόρυξης. Και αν τα προϊόντα αυτής της δραστηριότητας χρηματοδοτούν εκ των υστέρων της σειράξεις αυτές. Αυτό έχει τεράστιες συνέπειες για εκατομμύρια ανθρώπων κατοίκων των περιοχών αυτών, στην Αφρική κυρίως ιδιαίτερα δε στην κεντρική περιοχή των μεγάλων λιμνών. Εξετάζει λοιπόν και εκτιμά η έκθεση αυτή το ότι γίνεται σε τέσσερις καταγεγραμμένες περιοχές συγκρούσεων πιο συγκεκριμένα. Ε, τα προβλήματα που δημιουργούνται από την παραγωγή των ορυκτών αυτών είναι πάρα πολύ σοβαρά. Προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι αιτίες, ποιοι είναι οι λόγοι οι οποίοι τροφοδοτούν και προκαλούν αυτές τις σειράξεις. Και ταυτόχρονα να δούμε τι λύσεις μπορούμε να βρούμε. Θα πρέπει για να το κάνουμε αυτό βέβαια να δούμε ποιες είναι οι αιτίες. Έλλειψη κλίματος ασφαλείας, έλλειψη κυβερνητικών σταθερών δομών, έλλειψη υποδομών, γενικότερη διαφθορά ή άλλα πλαίσια. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να λάβουμε υπόψη μας δράσεις και σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο στα πλαίσια των εμπορικών δραστηριοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς αυτών των ουσιών όπως ο κασίτερος, το βολφράμιο και το ταντάλιο εισάγει το 35% της συνολικής παραγωγής αυτών των τριών μετάλλων και υπάρχουν και χώρες άμεσες εισαγωγής αυτού του τύπου των μετάλλων. Είμαστε υπεύθυνοι λοιπόν για την εμπορία των συγκεκριμένων αυτών προϊόντων και θα πρέπει ακριβώς να τεθεί το θέμα εδώ της δέουσας ε, επιμέλειας της δέουσας επιμέλειας και για τη συνεργασία μας, την συνεργασία μας με τις χώρες αυτές οι οποίες ε, ε, παίρνουν μέρος σε αυτού του είδους τις εμπορικές συναλλαγές. Συγκεκριμένη περίπτωση τις εισαγωγές και να δούμε τι σχέσεις έχουν βέβαια αυτές οι εξορίξεις, οι δραστηριότητες με τις πολεμικές δραστηριότητες και με, ε, και με τα φαινόμενα διαφθοράς. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο να επιβάλλουμε ένα εμπάργο στα προϊόντα αυτής της ζώνης όπως τις μεγάλες λίμνες, αλλά αυτό θα προκαλέσει το ανάποδο αποτέλεσμα γιατί κάποιες χώρες θα προχωρήσουν στην εκμετάλλευση αυτή χωρίς έλεγχο και ανεξάρτητα. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι στα πλαίσια της νομοδότησης για αυτό το κανονισμό έχει σημασία η λεγόμενη αυτοπιστοποίηση των εισαγωγών αυτών, λαμβάνοντας υπόψη το τι συμβαίνει στις χώρες αυτές που είναι σε περιοχές ε, συγκρούσεων και αναφέρομαι κυρίως στην ε, ε, δημοκρατία του Κονγκό. Είναι σαφές να συνειδητοποιούμε ότι γενικά στο σύνολο της διαδικασίας αυτής μπορεί κανείς να παρέμβει και ακριβώς ε, μέσω ακριβώς της δέουσας επιμέλειας, ε, της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας ε, να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις διαδικασίες αυτές. Είμαι λοιπόν στην διάθεσή σας και θα συνεργαστώ και με τους, σκιώδους, τους σκιώδεις εισηγητές που θα ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σαρτζεντίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρέπει να είμαι στον τριμερή διάλογο για την καταπολέμηση του ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος. Τον Φεβρουάριο η Επιτροπή Ανάπτυξης πέρασε μια, ψήφισε μια έκθεση την οποία εγώ κατέθεσα για την υπεύθυνη ε, χρήση και εμπορία των ε, προϊόντων εξόριξης και τέθηκαν κάποια βασικά κριτήρια ε, για την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα κριτήρια αυτά ήσαν επακριβέστατα και υπήρξε μια καλή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο που τη στήριξε, τα περισσότερα κόμματα τη στήριξαν την πρόταση. Τώρα η πρόταση την οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ε, δεν ευθυγραμμίζεται με αυτά τα οποία είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις υπεύθυνε προμήθειες προϊόντων. Οι πράσινοι πιστεύουν ότι στην ουσία έχουμε να κάνουμε με μια εθελοντική αυτορύθμιση πρώτων υλών γιατί δεν εμπλέκονται όλες έτσι και αλλιώ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λόγω του ότι η ρύθμιση αυτή ε, στηρίζεται στην εθελοντική συμμετοχή. Δεν επιβάλλουμε στις επιχειρήσεις κάτι που θα θεωρηθεί ιδιαίτερα γραφειοκρατικό. Μιλάμε μόνο για τις πρώτες ύλε, όπου η οπληψηφία των πρώτων υλών που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πρώτες ύλε, είναι επεξεργασμένα καγαθά, υπολογιστές, iPads, ε, κινητά τηλέφωνα και τα οποία μάλιστα παράγονται όχι στην Ευρώπη αλλά κυρίως στην Νοτιοανατολική Ασία και πιο συγκεκριμένα στην Κίνα. Εάν όμως θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πραγματική ζήτηση για τα ορυκτά αυτά τα μέταλλα τα οποία προέρχονται σε περιοχές όπου έχουν αποτύχει τα κράτη ε, στον οποίο την επικράτεια γίνεται η εξόριξη αυτή, τότε θα πρέπει να βρούμε ένα νέο σύστημα όπου όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδείξουν αυτή την δέουσα επιμέλεια. Αν δεν το επιβάλλουμε αυτό τότε δεν προσθέτουμε τίποτα, δεν διορθώνουμε τίποτα ε, στην, ε, στον Αμερικανικό νόμο Dot Frank το οποίο περιορίζεται σε ε, εισηγμένες επιχειρήσεις και όχι σε επιχειρήσεις οι οποίες ε, ασχολούνται ε, με, με τη δημοκρατία του Κονγκό και με τις περιβάλλουσες περιφέρειες σε αυτήν. Νομίζω ότι μάλιστα οι περιοχές αυτές είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Ακούω πάρα πολλά παράπονα για τον νόμο Dodd Frank, για τη νομική ρύθμιση Dodd Frank που στην ουσία επιβάλλει de facto embargo. Εγώ το αμφισβητώ αυτό. Το 2010 όταν οι Ηνωμένε Πολιτείες προώθησαν τη συγκεκριμένη νομοθετική ε, ρύθμιση χωρίς τις λεπτομέρειες, τη γενική ιδέα. Οι Αμερικανικές επιχειρήσεις αποχώρησαν γιατί είπαν ότι καλύτερα να φυλάγονται. Αλλά τώρα φαίνεται ότι επανέρχονται οι Αμερικανικές επιχειρήσεις και αρχίζουν πάλι να επανέρχονται ε, και όπως είπα να προμηθεύονται από το Ανατολικό Κονγκό προϊόντα. Και μάλιστα ο πρόεδρος ο Καμπίλα έχει επιβάλει στη δική του χώρα ε, μια απαγόρευση εξαγωγών κανονικά στην χώρα του για τα προϊόντα αυτά. Αυτά λοιπόν έχουν οδηγήσει σε μία μείωση στις εξαγωγές, αλλά είδαμε όμως μία αύξηση στις εξαγωγές τελικά από το ανατολικό κομμάτι, το ανεξέλεγκτο του DRC, της Δημοκρατίας του Κονγκό και οι επιχειρήσεις αυτές φαίνονται ότι επανέρχονται. Οπότε είναι κρίσιμο για να γίνουν τα επόμενα αυτά βήματα και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να συμπεριληφθούν, ιδιαίτερα αυτές που προωθούν τα λεγόμενα καταναλωτικά προϊόντα και αν δεν μιλάμε για την εμπορία των επεξεργασμένων προϊόντων, τότε δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για το σύνολο των καταναλωτικών προϊόντων. Ε, το ποσό, το, το, ο όγκος μάλλον των προϊόντων αυτών των προς επίπεδο πρώτης ύλη, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επεξεργασμένων προϊόντων στην Ευρώπη, είναι πάρα πολύ ε, μικρό. Απαιτείται λοιπόν αν θέλουμε να επηρεάσουμε την κατάσταση στο Κονγκό να, ε, ε, να ενημερώσουμε τον Ευρωπαίο καταναλωτή, κάτι το οποίο δεν κάνει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μια τελευταία παρατήρηση Πρόεδρε. Η συγκεκριμένη πρόταση την οποία η Επιτροπή ΙΤΑ σε αυτή τη φάση συζητά και προσπαθεί να επηρεάσει συνοδεύεται από μια ανακοίνωση. Μια ανακοίνωση η οποία περιλαμβάνει τα λεγόμενα συνοδευτικά μέτρα. Δεν έχουμε όμως ακόμα πάρα πολλές πληροφορίες γι' αυτό. Από ό,τι φαίνεται το πρόγραμμα και στη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ και στην Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει λοιπόν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτές, γιατί αυτό το οποίο πράγματι θέλουμε να έχουμε στη διάθεσή μας είναι κάποια αποτελεσματικά μέτρα, κάποια ασφαλή μέτρα και για τις διεθνείς επιχειρήσεις και για τις τοπικές επιχειρήσεις σε μια χώρα σαν τη Δημοκρατία του Κονκό να μπορούν να επενδύουν και να αγοράζουν προϊόντα γιατί αλλιώς θα κάνουμε μια ρύθμιση μονομερή στην Ευρώπη, στην ουσία δηλαδή ε, θα επιβάλλουμε μια απαγόρευση εισαγωγής ε, χωρίς να διορθώσουμε τίποτα επιτόπου. ιδιαίτερα για τα μέταλλα αυτά από τις δύσκολες περιοχές. Απαιτείται το σύστημα να μην είναι εθελοντικό, να είναι υποχρεωτικό και να υπάρχουν σοβαρά συνοδευτικά μέτρα. Ευχαριστώ. Περνάμε στις άλλες ε, πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Νόρπερτ. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ τον ΣΕΠ, ο οποίος δεν μπορούσε να είναι σήμερα, εδώ. Καλά, μου αρέσει και επικροτώ την προσέγγιση του εισηγητή. Εμείς πιστεύουμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αδύναμη και δεν έρεται στα επίπεδα των άλλων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό προσβλέπουμε και στην Επιτροπή ΝΤΕΒ και στην Επιτροπή ΙΝΤΑ να ε, συνεργαστούμε ώστε να είναι πιο φιλική προς την ανάπτυξη η πρόταση αυτή που πρέπει να είναι όπως και το σύστημα αυτό ε, πιστοποίησης ε, να είναι υποχρεωτικό και όχι εθελοντικό. Έτσι θα ευθυγραμμιστούμε με τις αγορές στις ΗΠΑ και θα ανταποκριθούμε και στις εξελίξεις της κινέζικης αγοράς επειδή έχουμε εμπορικά ε, συμφέροντα, δεν θέλουμε να υπονομευθούν από το εμπόριο μεταλλευμάτων από περιοχές ε, συγκρούσεων. Δεν μπορούμε να έχουμε χαμηλότερα πρότυπα από αυτά των ΙΠΑ και της Κίνας. Ε, επίσης, το πεδίο εφαρμογή θα πρέπει να διευρυνθεί, γιατί δεν είναι επαρκή τα μεταλλεύματα τα οποία περιλαμβάνονται θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο κατάλογος όλων των ε, κρίσιμων μεταλλευμάτων στη μελλοντική νομοθεσία για να μην έχουμε αποσταθεροποίηση κάποιων αγορών ε, ή εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον και για να μην ε, μένει εκτός νομοθεσίας καμία περιοχή συγκρούσεων στο μέλλον. Πρέπει λοιπόν η περιοχή συγκρούσεων ως όρος να προσδιοριστεί πολύ καλύτερα όχι όμω να περιορίσουμε γεωγραφικά το πεδίο εφαρμογή λέγοντα ε, περιοχή μεγάλων λιμνών. Έτσι θα μπορούμε να τοποκριθούμε σε νέε αναδιόμενες συγκρούσει Και μάλιστα τάχιστα τέλος. Δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο τους, πρωτογενεί πρωτογενείς αγωγείς ε, πρώτων αλλά και όλες τις ε, επιχειρήσεις που εισάγουν τελικά προϊόντα ή, ή μη επεξεργαμένα, τα οποία περιλαμβάνουν αυτές τις ουσίες για το χρυσό και πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ε, και οι όροι για την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, υποσημείωση. Θα πρέπει προτάσεις να συνοδεύονται από μέτρα που θα παρέχουν υποστήριξη, κίνητρα και ένα βελτιωμένο πλαίσιο για την νόμη εκμετάλλευση και την διατεχνική ε, εκμετάλλευση αυτών των μεταλλευμάτων θα πρέπει να αποτρέψουμε και περαιτέρω συγκρούσεις και βέβαια και την υπομνόμευση του αναπτυξιακού έργου. Είναι φιλόδοξη η ατζέντα. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για αυτό το νομοθέτημα. Ελπίζουμε να αποδώσει και για μας αλλά και για τις χώρες των αψόμενων, των κόσμου τα μέγιστα. Ευχαριστώ. ECR εκπρόσωπος, ο κύριος Ντέβα. Ευχαριστώ. Άκουσα προσεκτικά τα όσα είπε η κυρία Σαρσεντίνη και ο κύριος Νόισερ και συμφωνώ απολύτως με όλα αυτά που είπαν και οι δύο. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει κανονισμός ή κανένας έλεγχος αν δεν είναι υποχρεωτικός. Τώρα έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα για τα διαμάντια που προέρχονται από αυτές τις περιοχές. Χρειάστηκε πάρα πολύ καιρός για να έρθει αυτή η νομοθεσία κάθε ε, πολύτιμος λίθος που μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχεται για να μην έρχεται από διαμαντορυχείο που ε, είναι στα χέρια ε, πολεμάρχων. Χιλιάδες χιλιάδων ανδρών, γυναικών και παιδιών έχουν χάσει τη ζωή τους, ιδιαίτερα στην Αφρική. Γιατί υπάρχουν κάποιοι πάρα πολύ άπλιστοι άνθρωποι και έχουν εκμεταλλευτεί διαφορές και εδαφικές και φιλετικές για να κάνουν ένα πιάτσικο εκεί στις χώρες αυτές. Αν γινόταν κάτι τέτοιο λοιπόν και έφτανε τέτοιο διαμάντι στις Βρυξέλλες, ε, δεν θα ήταν επιτρεπτό. Γιατί να γίνεται αλλού. Λοιπόν, αντλώντας ε, αυτά τα διδάγματα από την εμπειρία ε, της διαδικασίας του Κίμπερλι, για ποιο λόγο να μην έχουμε την ίδια μεταχείριση με τα διαμάντια και στα μεταλλεύματα. Αφήστε που και τα διαμάντια είναι μεταλλεύματα. ή και τα μεταλλεύματα διαμάντια. Γιατί να κάνουμε γραφειοκρατικές ανοησίες. Υπάρχουν οι βέλτιστες πρακτικές αυτές και θα πρέπει να πούμε ε, στην κοινότητα αυτή ότι για να έχουμε ένα κανονισμό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός, αλλιώς τι να το κάνουμε. Θα ε, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Να φτιάξει ένα μισθοφορικό στρατό, να πάει να σκάβει, ε, να, να κλέβει το χρυσάφι του κόσμου. Ε, κάπως έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με το σωστό τρόπο και όπως είπε και ο συγητής, θα είμαστε τελικά περήφανοι για αυτή την νομοθεσία, εάν περάσει με το σωστό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από την Άλντε, Κάθε και μετά η Λόλα από την ΚΟΕ. Εδώ και ένα χρόνο είχα τη δυνατότητα μαζί με την Τζούδιθ να επισκεφθώ τη Ρουάντα, τον Μπουρούντι και τη Δημοκρατία του Κογο και είδα ε, την εξόριξη αυτών των μετάλλων. Είδα τον κόσμο να ε, μπαίνει μέσα στις ε, τρύπες με, με, με κομμάτια μέταλλο από παλιούς τράκτορες και όχι ούτε καν με φτιάρια αλλά εν πάση περιπτώσει είδαμε τις απαράδεκτες συνθήκες και είδαμε τα μέταλλα αυτά να εξορίσονται και ξέρουμε ότι χάνονται τα μισά δεξιά και αριστερά πριν φτάσουν στον τελικό παραλήπτη. Ε, συνεργαστήκαμε επίσης και με μια επιχείρηση αρκετά ανεξάρτητη στην Ρουάντα και μας είπε και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε και για την έκθεση ότι καθιστώντας πιο αυστηρά τα μέτρα γύρω από την κατάσταση αυτής της ε, ζώνες σύραξης ε, και επηρεάζοντα έτσι το ευπόλυτο των ε, πρώτων αυτών υλών η Αυστραλία και κάποια άλλη παραγωγή των μετάλλων στην ουσία θα δουν οι τιμές των προϊόντων τους να πέφτουν πάρα πολύ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει τις συμφωνίες που έχουμε. Γιατί θα πλημμυρίσουν τα προϊόντα αυτά της Δημοκρατίας του Κονγκό ε, τις κοινοτικές και διεθνείς αγορές με συνέπειες ε, για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Πρέπει να καταστήσουμε τα ορυχεία αυτά ασφαλέστερα για αυτούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκεί, ε, να τα καταστήσουμε πιο ελκυστικά σε επίπεδο αποδοτικότητας, αλλά θα επηρεάσουμε αρνητικά τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου. Said, uh, why can't we use the same traceability of diamonds? Diamonds come directly to the uh, EU and are cut. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα επηρεάσει αυστηρά την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις υπόλοιπες χώρες παραγωγούς. Και ε, θα δούμε ότι ε, έτσι και αλλιώ τα προϊόντα αυτά πηγαίνουν πρώτα σε άλλες χώρες και έρχονται σε εμά υπό τη μορφή κινητών τηλεφώνων ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω λοιπόν ότι σαν Επιτροπή Ανάπτυξης θα πρέπει να τονίσουμε ε, και τη σημασία της παραγωγής σε διάφορες χώρες και της προτιστέμενης αξίας. Δηλαδή είναι παράλογο να επιμένουμε οι χώρες αυτές να εξάγουν αυστηρά τις πρώτες ύλες. Πρέπει να υπάρχει προστιθέμενη αξία. Αυτό θα δώσει ικανότητες, δυνατότητες επεξεργασίας και επιπλέον χρήματα απόδοση και ανάπτυξη. Γιατί έτσι και αλλιώς βλέπουμε ότι τα επεξεργασμένα προϊόντα ε, γίνονται ε, πιο ευνοϊκά δεκτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν προϊόντα εισαγωγής από ότι ε, ο πρώτος, οι πρώτες ύλες. Τώρα για τα προϊόντα λαιλασίας. Πράγματι και οι Ηνωμένε Πολιτείε παλιότερα, αλλά τώρα η Κίνα λαιλατούν σε επίπεδο πρώτων υλών την Αφρική. Θα πρέπει εμείς να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να έχουν μια ασφαλή αγορά, να είναι ανοιχνεύσιμα τα προϊόντα αυτά, να γνωρίζουμε ότι δεν εμπλέκονται εγκληματικές δραστηριότητες, ότι υπάρχει υψηλή προστιθέμενη αξία και εν πάση περιπτώσει να είναι χώρες οι οποίες ε, να μην εξαρτώνται από την βοήθεια των ξένων χωρών αλλά να μπορέσουν μόνες τους να παράγουν πλούτο. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος ο οποίος θα ήθελε το λόγο και θα θέσω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις και εγώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διάβασα και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακούσαμε και τη συζήτηση που προηγήθηκε και πράγματι υπάρχει συνένεση στο ότι κάτι θα πρέπει να υπάρξει τώρα για το αν θα είναι θελοντικό ή ε, υποχρεωτικό το καθεστώς θα δούμε. Αυτό το οποίο εσείς πραγματικά προτείνετε είναι ένα πρόγραμμα κατευθυντηρίων γραμμών έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να προσυπογράψουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις από το 2010. Στην ουσία δηλαδή ε, εσείς ζητάτε ένα ε, προαιρετικό σύστημα ετικετοθεσίας σε εισαγωγικά των προϊόντων. Αλλά οι αξιολογήσεις που είχατε κάνει εσείς ε, το 2010 ε, δεν έχουν ε, φέρει στην επιφάνεια κάποια θετικά βήματα, κάποια πρόοδο. Τι έχει αλλάξει από το status quo αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας είναι λίγο ξεπερασμένα. Τι καινούργια πράγματα και τι έχει αλλάξει. Η Σαρτζεντίνη επίση θέλει να μάθει τι γίνεται ακριβώς και με τα συνοδευτικά μέτρα. Είχατε πει το Μάρτιο ότι θα υπάρξει ένα πακέτο μέτρων. Πού είναι αυτό το πακέτο. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να πάρει το λόγο κάποιος από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου ή μόνο από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. Αλλά οι προτάσεις αυτά για τα συγκεκριμένα μέτρα σε ποια φάση βρίσκονται. Ε, πόσες επιχειρήσεις έχουν προσυπογράψει μέχρι τώρα. Ε, η πρότασή σας ε, συνίσταται στο να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα και κάθε κράτος μέλος θα έχει μια υπηρεσία που θα παρακολουθεί την σωστή εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων. Δεν θα υπάρχει κάτι σε, σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο και οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες να μας πούν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν τις συγκεκριμένες, ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αυτών. Και τέλος, από ό,τι φαίνεται, σχετικά πάντα με τις πρώτες ύλε και την συζήτηση ανάμεσα στις πρώτες ύλε και τα επεξεργασμένα προϊόντα. Πράγματι προωθείται η ιδέα της προτίμησης των επεξεργασμένων προϊόντων Ξέρω ότι οι επιχειρήσεις αυτές προτιμούν και θα επιλέξουν την προαιρετική λύση, αλλά το θέμα είναι να τις πείσουμε να υπακούσουν στις ρυθμίσεις. Μήπως πρέπει τελικά να προτείνουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο έχουν εφαρμόσει οι Ηνωμένε Πολιτείε. Είχε γίνει μια τέτοια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχάς, αλλά από ό,τι φαίνεται απερίφθη στο τέλος της διαδικασίας. Μήπως πρέπει να έρθετε σε επαφή με τους Αμερικανούς νομοθέτες και να μπορέσετε να κατανοήσετε ακριβώς το τι συμβαίνει στις Ηνωμένε Πολιτείε με αυτό. Ε, το γραφείο μας στην Ουάσιγκτον μπορεί να μας βοηθήσει να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει με την εφαρμογή του ε, νομοσχεδίου Frank Dot. Λοιπόν, στην περίπτωση που εμείς ε, ασχοληθούμε μόνο με τους εισαγωγείς, εδώ όμως βλέπουμε ότι οι περισσότεροι αυτοί που επεξεργάζονται και προχωρούν στην τήξη των μετάλλων αυτών είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε πώς θα επηρεάσουμε θετικά την κατάσταση. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω, κάποιος άλλος δεν θέλει το λόγο, οπότε θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου. Yes, uh, good afternoon to all. Thank you, Chair. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. ετέθησαν διάφορα ερωτήματα, αλλά θα ήθελα αν μου επιτρέπετε να σας υπενθυμίσω σε συντομία το ιστορικό της πρότασης, ε, ποια είναι τα βασικά της χαρακτηριστικά και όταν περιγράψω αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά, ίσως απαντηθούν και ορισμένα από τα ερωτήματα. Λοιπόν, η πρόταση αυτή ήλθε μετά από πολύ προπαρασκευαστική δουλειά διοργανώθηκε διαβούλευση, είχαμε μια μελέτη αντικτύπου, προπαρασκευαστική φάση διάρκεια ενός έτους και μετά υποβάλαμε αυτή την πρόταση το Μάρτιο του 2014 συγκεκριμένα. Και πρόκειται περί πακέτου το σχέδιο κανονισμού για αυτό το σύστημα αυτοπιστοποίησης για τη δέωση επιμέλεια για τους ε, εισαγωγείς κασιτέρου, Βολφραμίου, τανταλίου και χρυσού, μαζί με μια κοινή ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπα της εκπροσώπου, που αφορούσε τη ευρύτερη πτυχή, δηλαδή της υπεύθυνη εξόρισης μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου. Όλα αυτά έγιναν σε ανταπόκριση εκκλήσεων και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφέρθηκε η κυρία Σαρχεντίνη σε ορισμένα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αυτό το θέμα. Και ο στόχος μας μεταξύ άλλων ήταν βασιζόμενοι στις διεθνείς προσπάθειες και στην αναδυόμενη συνένεση που υπάρχει γύρω από αυτές τις γραμμές του ΩΣΑ να κάνουμε ένα βήμα περαιτέρω. Πρέπει βέβαια να συμφωνήσουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο δεσμευτικό νομικό πλαίσιο σε διεθνές επίπεδο για αυτό το ζήτημα. Έγινε αναφορά στα διαμάντια και στη δικασία Κίμπερλι. Ε, βέβαια, εδώ έχουμε ένα διαφορετικό πλαίσιο, υπό την έννοια ότι είναι πιο στέρεο Συμπαγέ το πλαίσιο για την υιοθέτηση κάποιων κανόνων σε αυτό το τομέα των διαματιών. Αν τώρα θέλουμε να κάνουμε σύγκριση με άλλα συστήματα υφιστάμενα, για το ξύλο, για τα διαμάντια, για το ξύλο ξέρω υπάρχει ένας νέος κανονισμός, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι εδώ μιλούμε για προϊόντα με πολύ μακρά αλυσίδα εφοδιασμού. 7, 8, 9 χρόνια. Άρα η δέωσα επιμέλεια γίνεται πιο πολύπλοκη διαδικασία και η παρακολούθηση της αλυσίδας εφοδιάς μου βέβαια. Έχουμε και τρεις συμπληρωματικούς στόχους που υπηρετούν την παρουσίαση αυτής της πρότασης. Υπάρχουν ε, στόχοι που είναι συμπληρωματικοί όπως είπαμε μεταξύ τους. Πρώτο, εξόριξη μεταλλευμάτων και χρηματοδότηση συγκρούσεων. Αυτός ε, ο δεσμός πρέπει να σπάσει. Αυτή είναι η πρώτη ε, μέρημνά μας. Επίσης να ελέγξουμε τι γίνεται επιτροπές συγκρούσεων, ε, περιοχές συγκρούσεων, να μην έχουμε εξαγωγή μεταλλήματων από αυτές τις περιοχές και να δούμε συμμόρφωση, αν υπάρχει συμμόρφωση των κρατών μελών προς τα συστήματα της δέωσας επιμέλειας και αναφερθήκατε και στο νόμο το ΤΡΑΚ που ισχύει στο, στην περίπτωση των Πολιτειών. Uh, uh, Υπάρχει λοιπόν η πρόλεψη για αυτό το σύστημα αυτοπιστοποίησης των υπεύθυνων εξαγωγέων και ε, εισαγωγέων που προαιρετικά εντάσσονται αυτό στο σύστημα προβλέπονται υποχρεώσει δέωσης επιμέλειας. Υπάρχουν φορείς ε, οι οποίοι θα αξιολογούν τη συμμόρφωση και ενδέχεται και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους να διενεργεί ελέγχους. Τέσσερα είναι τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του σχεδίου κανονισμού. Και θέλω να τα επαναλάβω γιατί νομίζω θα απαντήσουν πολλά από τα ερωτήματά σας. Πρώτο, γεωγραφικό πεδίο εφαρμογή, γεωγραφικό εύρος κανονισμού. Είναι ευρύ το γεωγραφικό αυτό πεδίο. Θέλουμε να καλύψουμε όλες τις περιοχές συγκρούσεων και ψηλού κινδύνου. Να μην περιοριστούμε μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή που είναι η προσέγγιση της νομοθεσίας Dodd Frank στη ΣΥΠΑ. Δεύτερο, σε σχέση με τα προϊόντα. Έχουμε αυτά τα τρία μεταλλεύματα συν το χρυσό, Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ έχουν αναπτύξει ε, με διάφορα παραρτήματα ε, τις σχετικές διατάξεις. Μοιάζουν με τη νομοθεσία Dodd Frank. Τρίτον, τρίτη πτυχή. Το επίπεδο της αλυσίδας ε, εφοδιασμού που εμείς προτείνουμε να γίνει παρέμβαση. Δεν προτείνουμε να έχουμε παρέμβαση κατάντι, downstream, όπως προτείνω με τη Dot Φρανκ, αλλά στο μέσο της όλης διαδικασίας, στο μέσο της αλυσίδας, ε, στο επίπεδο της επεξεργασίας. Γιατί εκεί είναι το κρίσιμο, κρίσιμο σκόμπο στην αλυσίδα. Και πρέπει να συλλεγούν πληροφορίες σε αυτό το στάδιο για σε επόμενα στάδια της διαδικασίας η συλλογή των αυτών των πληροφοριών δεν μπορεί να γίνει. Επίσης, στο πλαίσιο της ε, διαδικασίας διαβούλευσης ακούσαμε πολλές εταιρείε ε, που ε, αφορά και η εφαρμογή της Αμερικανικής νομοθεσίας να μας λένε ότι δεν έχουν αρκετές πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις ε, και επεξεργασίας αυτών των μεταλλευμάτων. Είναι μικρή κλίμακα. Μιλάμε για 400-500 τέτοιους ε, απασχολούμενους που κάνουν την τήξη και την επεξεργασία αυτών των μεταλλευμάτων. Αυτό είναι το επίπεδο που θεωρούμε ότι πρέπει να παρέμβουμε και οι πληροφορίες που θα συλλέξουμε σε αυτό το επίπεδο, αυτό θα είναι χρήσιμο για τις κατάντι επιχειρήσεις που όπως είπατε έχουν ε, υποχρέωση δυνάμει του συστήματος Dot Frank να φέρουν σε πέρα σε τις διατάξεις δέουσας επιμέλειας. Πρέπει να έχουμε λοιπόν αυτές τις πληροφορίες. Και αυτό εννοούσα όταν είπα συμπληρωματικότητα με την νομοθεσία Dot Frank. Τώρα, η νομοθεσία μας θα ισχύει στους εισαγωγείς των τεσσάρων αυτών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μικρά, μικρό σχετικά αριθμητικά ο πληθυσμός αυτός. Υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στους 400 ε, οι εισαγωγείς ε, των προϊόντων αυτών. Επίσης, το σχέδιο κανονισμού περιλαμβάνει διατάξεις που αναφέρουν ότι βάσει των συλλεγισών πληροφοριών μέσω αυτού του συστήματος αυτοπιστοποίησης ε, δημοσιεύεται ετησίως ένας κατάλογος των ε, εγκαταστάσεων τήξης και επεξεργασίας μεταλλευμάτων μεταξύ των οποίων και αυτών που κάνουν αυτή τη δέωση και μπορούν να πιστοποιήσουν ότι είναι καθαρά τα μετάλλευματά του, τα προϊόντα του. Ενημερώνεται, επικαιροποιείται το κατάλογος αυτός. Και αν ασκηθεί πίεση και από εσά μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο αυτή η διαδικασία. και να συμβουλεύονται περισσότερο τον κατάλογο αυτό. Άκουσα τι είπατε για τις κατευθύνες γραμμές ε, του ΩΣΑ. Πιστεύω ότι θα ασκηθεί μια πίεση από μοτίμους αν ε, έχουμε αυτή μικρή ομάδα που θα κληθεί να εφαρμόσει το σύστημα. Και τώρα έρχομαι σε κάτι που άκουσα σε πολλές παρεμβάσεις. Ήτι στον εθελούσο χαρακτήρα αυτής της πρότασης έναντι υποχρεωτικού ε, δυνητικά χαρακτήρα αυτής της πρότασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να είναι εθελοντικό το σύστημα. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αποφύγουμε καταστάσεις όπου θα υπήρχε κίνδυνος κάποιες πληροφορίες να πάψουν να δραστηριοποιούνται σε περιοχές κινδύνου ή συγκρούσεων, κάτι που έχουμε ήδη παρατηρήσει στο πλαίσιο της νομοθεσίας Dot Frank για την περιοχή των μεγάλων λιμνών συγκεκριμένα μιλώ. Εμείς παρακολουθούμε και διαβάζουμε και πολύ προσεκτικά τις εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων ε, του ΟΣΑ και του ΟΗΕ. Είναι εκθέσεις οι οποίες δημοσιεύονται ε, σε αιτήσια βάση και αναφέρουν ότι υπάρχει αύξηση στο λαθρεμπόριο και μείωση της παραγωγής. Σημαντική μείωση και των εισόδων βέβαια σημαίνει αυτό για τις ε, αρχές που θα μπορούσαν να έχουν αρκετά έσοδα από τις εξαγωγές αυτών των προϊόντων. Επίσης είδαμε από ορισμένε επιχειρήσεις, ε, αρκετές στον αριθμό, να ζητούν από τις προμηθευτές τους ε, να μην αγοράζουν από αυτές τις περιοχές. Υπάρχει βέβαια και δίκαιο εμπόριο σε περιοχές συγκρούσεων όμως η συνολική εικόνα είναι ανησυχητική. Βλέπουμε αυτό το κίνδυνο απεμπλοκής, αν μπορώ να το πω έτσι, και ο κίνδυνος αυτός είναι πραγματικός. Θέλουμε να αποφύγουμε να εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές. Άλλωστε το πεδίο εφαρμογή ε, είναι ευρύ και αν πάμε σε ένα υποχρεωτικό σύστημα θα υπήρχε ο κίνδυνος παρέμβασης σε περιβάλλοντα που είναι ρευστά, σταθή, εύθραυστα και εκεί να δημιουργηθεί πάλι αυτό το πρόβλημα της απομάκρυσης, απεμπλοκής κάποιων επιχειρήσεων. Πώς μπορεί να παραχθεί ζήτηση είναι ένα θέμα, αλλά δεν είναι το μόνο μέλημά μας. Πολλοί είναι οι λόγοι λοιπόν για τους οποίους θεωρούμε ότι το εθελοντικό σύστημα είναι προτιμότερο του υποχρεωτικού. Βέβαια η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχει εκπονηθεί με πολύ μεγάλη προσοχή και επιμέλεια. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε το σύστημα επαρκώς και γι' αυτό στην πρότασή μας αναφέρουμε ότι θα υπάρξει μια αξιολόγηση μετά από τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής αυτού του συστήματος. Και ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αξιολόγηση αυτή διατυπώσει προτάσεις και ίσως εισαγάγει και κάποια υποχρεωτικά στοιχεία σε αυτό το σύστημα. Είναι σαφές ότι όταν κάνουμε την αξιολόγηση θα λάβουμε υπόψη μας όλος ιδιαίτερος ε, το πόσο χρησιμοποιείται αυτό το σύστημα από τους εισαγωγείς. Τώρα, και πάλι, η πρόταση συνοδεύεται από μία ανακοίνωση για τα συνοδευτικά μέτρα. Ένα από τα συνοδευτικά αυτά μέτρα που έχει ιδιαίτερη σημασία πιστεύω για να αντιμετωπίσουμε και το άλλο ζήτημα που άκουσα από πολλά μέλη που είναι οι πρώτη ύλε σε σχέση με το βιομηχανικό τελικό προϊόν. Ένα σημαντικό κίνητρο έχει να κάνει με τις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες. Και στην ανακοίνωση δηλώσαμε ότι θα δοθούν κίνητρα με ρήτρες επιδόσεων στις δημόσιες συμβάσεις που θα συνάπτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις επιτρέπει τέτοιες ρήτρες επιδόσεων. Η πιο πρόσφατη εκδοχή που εγκρίθηκε το προβλέπει αυτό Οπότε έχουμε αναλάβει τη δέσμευση ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλαμβάνουμε τέτοιες ρήτρε στις συμβάσεις μας για τις δημόσιες προμήθειες και έχουμε απευθύνει έκκληση και στα άλλα θεσμικά όργανα αλλά και στα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν αντίστοιχες ρήτρε στις δικές τους συμβάσεις για τις δημόσιες προμήθειες. Αυτό τι σημαίνει. Για να κερδίσει ένα διαγωνισμό και ένα συμβόλαιο μια εταιρεία θα πρέπει να αποδείξει ε, μέσω ε, διαδικασιών δέουσας επιμέλειας ότι έχει ελέγξει την ειχνηλασιμότητα των προϊόντων και έχει επιδείξει αυτή την δέουσα επιμέλεια. Είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο και αν θέλετε θα συμπεριλάβει τελικά σε όλη αυτή τη διαδικασία και τα τελικά βιομηχανικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρε, και εσείς κάνατε κάποιες ερωτήσεις στο τέλος. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένες από τις ερωτήσεις σας. Ναι, σωστά ε, και αναφερθήκατε στην εφαρμογή από τα κράτη-μέλη ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση όλων αυτών και ποια είναι η συνήθις θεσμική ισορροπία ε, και πώς θα εφαρμοστεί δηλαδή η νομοθεσία θα γίνει με τρόπο ισόρροπο αυτό είναι απόκειται στα κράτη-μέλη και προβλέπεται από το σχέδιο κανονισμού. Βεβαίως γνωρίζουμε και εμείς ότι θα πρέπει να αποφύγουμε αποκλήσεις στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η νομοθεσία. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και την πρόθεση να εγκρίνουμε και να εκδώσουμε κατευθυντήριες γραμμές για να εξασφαλίσουμε την ομοιόμορφη ε, εφαρμογή της ε, κοινοτικής νομοθεσίας. Ρωτήσατε επίσης για τα συνοδευτικά μέτρα, ένα ανέφερα, το οποίο έχει να κάνει με τις δημόσιες συμβάσεις, υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, η παροχή βοήθειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικονομικής αλλά και τεχνικής στην ε, διεξαγωγή ε, κάποιων ελέγχων δέους επιμέλειας. Υπάρχει βέβαια και το θέμα του πολιτικού διαλόγου με τις τρίτες χώρες. και οι χώρες ε, του ΑΣΕ, του ΟΣΑ, συγγνώμη, ε, και ε, μιλήσατε και για τις προσπάθειες που κάνουν οι κινέζικες αρχές, που είναι πολύ νέα προσπάθεια αυτή και έγινε χάρη στην κοινή πίεση που ασκείται στις αρχές των τρίτων χωρών και μάλιστα χωρών όπως η Κίνα που έχουν πολλές ε, καταστάσεις στήξης και επεξεργασίας τέτοιων μετάλλων. Και η έγκριση της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κοινοτική νομοθεσία στον τομέα αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο επίσης ε, έδρασε καταλητικά για να κινητοποιηθούν περισσότερο οι κινέζικες αρχές. Βέβαια, πέρα από όλα αυτά και επιπλέον υπάρχουν και διατάξεις για αναπτυξιακή συνεργασία και τις έχουμε εκπονήσει ε, με τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΦΚΟ και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης με μεγάλη προσοχή και εδώ μπορώ να σας αναφέρω τις δράσεις που υπάρχουν ήδη σήμερα και το μέσον σταθερότητας Φερρυπίν όπου υποστηρίζουμε την εφαρμογή της... των αποφάσεων της Διεθνούς Διάσκεψης για την προστασία των πρώτων υλών της περιοχής των μεγάλων λιμνών για να αντιμετωπιστεί το θέμα της έφθραυστης αυτής περιοχής. Προωθούμε το θέμα της διαφάνειας στον τομέα της παραγωγής των μετάλλων αυτών και στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του ΟΣΑ για την δέουσα επιμέλεια στις εμπορικές δραστηριότητες, κάτι το οποίο έχει τύχει της πλήρου στήριξης από πλευρά της Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε επίσης και ε, την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών για τη χρήση της γης και την προστασία της γης σε περιοχές σειράξεων και θα βοηθήσουμε νομίζω μέσω της πλήρους συνεργασίας με τα υπόλοιπα διεθνή σώματα με το ενδεικτικό περιφερειακό πρόγραμμα σαν παράδειγμα για το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο για την Κεντρική Αφρική όπως και για το Παναφρικανικό Πρόγραμμα των ε, καθολικών αγαθών και των μελλοντικών προκλήσεων. Μελλοντικά ουσιαστικά προγράμματα τα οποία δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως τα οποία όμως θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε και οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση και από την άλλη υπηρεσία ότι χρειάζεται περαιτέρω συνεργασία με τους φορείς που τα προωθούν. Προσπαθούμε λοιπόν να ανταποκριθούμε με ένα ολοκληρωμένο τρόπο. Πρόεδρε, να τελειώσω με ένα τελευταίο θέμα. ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει κάποιο μέτρο το οποίο να είναι κατώτερο από το αντίστοιχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν το πιστεύουμε εμείς αυτό. Αντίθετα, το αμερικανικό σύστημα στην παρούσα φάση στην ουσία απλά επιβάλλει την υποχρέωση δημοσίευσης, δημοσιοποίησης. Αυτό το οποίο εμείς προτείνουμε είναι διαφορετικό. Εμείς προτείνουμε ένα σύστημα στα πλαίσια του οποίου αυτοί οι οποίοι εφαρμόζουν το, τις ρυθμίσεις αυτές θα πιεστούν από διάφορες πλευρές όπως από τις επιχειρήσεις τις συναλλασσόμενες, τους καταναλωτές να εφαρμόσουν το σύστημα. Και δεν περιοριζόμαστε στη δημοσιοποίηση αλλά δίδουμε εγγυήσει για το ότι εμείς τροφοδοτούμε την κοινοτική αγορά με προϊόντα σωστά σωστής προέλευσης. Έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές απόψεις λοιπόν. Δεν έχουμε παρμείνει εμείς μόνο στο σύστημα το αμερικανικό που επιμένει μόνο στο θέμα της διαφάνειας. Αντίθετα αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς είναι να αναλυφθεί δράση για αυτούς οι οποίοι εισάγουν προϊόντα από τις περιοχές αυτές. Λοιπόν αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να υπογραμμιστεί. Ελπίζω ότι έχω απαντήσει τα περισσότερα από τα θέματα που θέσατε. Αν όχι μπορώ να το κάνω αυτό είτε εδώ είτε διμερός με τα μέλη που θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ο κύριος Ντέβα θέλει κάτι να προσθέσει πριν δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της ε, ε, Ντέβε. Ακούσα πραγματικά ε, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας έδωσαν, τα οποία είναι δυστυχώς πολλά αλλά καθόλου πρακτικά, είναι πάρα πολύ περίπλοκα και υπερβολικά πολλά. Εσείς ε, στην ουσία θέλετε να ζητήσετε από αυτούς που προχωρούν στην τήξη των μετάλλων, που είναι 400 από αυτούς, να σας επικυρώσουν, να πιστοποιήσουν ότι τα προϊόντα τους δεν προέρχονται από περιοχές σειράξεων. Οι επιχειρήσεις αυτές ε, δεν ε, παίρνουν προϊόντα μόνο από ένα ορυχείο, ανακατεύουν προϊόντα διαφορετικής προέλευσης, εν πάση περιπτώσει, κάνουν μείγματα. Οπότε δεν μπορείτε εσείς να προχωρήσετε στη διαφοροποίηση ενός προϊόντος το οποίο έχει ε, περάσει από τη διαδικασία της τήξης αν προέρχεται από την Αφρική, από την Αυστραλία ε, ή από κάπου αλλού εν πάση περιπτώσει. Ε, ούτε μπορούμε να πούμε ότι ένα ποσοστό μπορεί να προέρχεται από μια περιοχή σύραξης. Λοιπόν, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες εδώ. Θα ήθελα όμως να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξής. Είπατε ότι κάνετε διαβουλεύσεις. Να μας πείτε γραπτά παρακαλώ, να ενημερώσετε την Πρόεδρό μας γραπτά για τις επιχειρήσεις οι οποίοι έκαναν, έδωσαν τα στοιχεία αυτά. Ποιοι είναι αυτοί. Καλώς. Πόσες επιχειρήσεις έχουν προϋπογράψει τις κατευθυντήριες γραμμές του ωσα. γιατί ήδη από το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προωθήσει τις ρυθμίσεις του ΩΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια εδώ και τέσσερα χρόνια. Πόσοι παίρνουν μέρος, σε πάση περιπτώσει. Είπατε επίσης ότι στα πλαίσια του Αμερικανικού συστήματος δεν μπορεί να ληφθούν μέτρα αν χρειαστεί στα πλαίσια των ρυθμίσεων αυτών. Οπότε ε, εσείς τι μπορείτε να κάνετε στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν θέλουν να πάρουν μέρος στο προαιρετικό σας σύστημα. Δεν ξέρω με ποιο βαθμό μπορείτε να ασκήσετε πίεση. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ αν μια επιχείρηση που παράγει το τηλέφωνο μου συμπεριλαμβάνεται ή όχι. Αναφερθήκατε στα οικονομικά κίνητρα στις επιχειρήσεις να υπακούν στις ρυθμίσεις αυτές. Πόσες λοιπόν έχουν χρησιμοποιήσει την προσφορά αυτή και υπάρχει ένας κατάλογος διαθέσιμος για τα μέλη του Κοινοβουλίου. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ. Ή μάλλον να δώσω τη δυνατότητα στην Trade να δώσει τις απαντήσεις τις πρώτες. Αν δεν έχετε απαντήσει σήμερα μπορείτε να μας τις στέλνετε γραπτά και θα τις μοιράσουμε εμείς στους συναδέλφους. Κάποιες από τις απαντήσεις τις έχουμε εδώ και θα σας στείλουμε και περισσότερες απαντήσεις γραπτά. Για την προηγούμενη παρέμβαση Η δυσκολία συλλογής πληροφοριών από τις εταιρείες που προχωρούν στην τήξη του προϊόντος είναι κάτι το ε, δεδομένο, είναι πολύ δύσκολο και αυτό το αντιμετωπίζει και η ρύθμιση DOT .frank. Θα πρέπει να προσπαθήσουν να ανοιχνεύσουν την αλυσίδα παραγωγής τους και προμήθειας για να μπορέσουν να δώσουν στοιχεία. Αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς στα πλαίσια του .frank Αυτό δείχνουν οι περισσότερες εκθέσεις. Λέγουν λοιπόν ότι η προμήθεια των προϊόντων τους είναι αόριστη, μη καθορισμένη. Και η διαβούλευση στην οποία εμεί είχαμε προχωρήσει δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες έμεσα εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις Dodd Frank λέγουν ότι το πιο δύσκολο στην αλυσίδα προμήθειας είναι ακριβώς ε, τι γίνεται σε επίπεδο επιχειρήσεων τήξης και επεξεργασίας. Οι επιχειρήσεις λοιπόν που χρειάζεται να υπακούν στις ρυθμίσεις Dodd-Frank ε, θα το κάνουν και με εμάς και εμείς θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το κομμάτι της ε, αλυσίδας προμήθειας όπου συλλέγουμε ακριβώς τις περισσότερες δυσκολίες για την ενημέρωση. Γι' αυτό λοιπόν επιμένουμε στη διαδικασία τήξης. Οι επιχειρήσεις τήξης αγοράζουν τα προϊόντα τους από διαφορετικά ορυχεία βέβαια, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις αυτές από πού προέρχεται η πρώτη ύλη. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πρώτη απάντηση στις παρατηρήσεις σας. και για τις παρατηρήσεις της Προέδρου. Η μελέτη την οποία έχουμε εμείς κάνει δείχνει ότι το 12% των επιχειρήσεων ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ. Τώρα για τον κατάλογο των επιχειρήσεων οι οποίες ήρθαν σε επαφή με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, νομίζω ότι αυτό δημοσιεύεται αν δεν κάνω λάθος, στη συνοδευτική τεκμηρίωση στα πλαίσια της έκθεσης για τη δημόσια διαβούλευση και τη μελέτη επιπτώσεων. Τώρα, αν δεν υπάρχουν ε, στοιχεία ενημέρωσης από πλευράς των εισαγωγέων, κοιτάξτε, είναι προαιρετικό το σύστημα. Ως εκ τούτου δεν έχουν την υποχρέωση να αυτοπιστοποιήσουν τους εαυτούς τους. Αλλά λόγω του μικρού τους αριθμού πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μια κάποια πίεση στους εισαγωγείς αυτούς έτσι ώστε να προμηθεύονται την πρωτεΐλη από την επεξεργασμένη πρωτεΐλη από πιστοποιημένες επιχειρήσεις τήξης και μονάδες επεξεργασίας που de facto θα δείξει ποιες είναι οι επιχειρήσεις αυτού του επίπεδου των οποίων τα προϊόντα είναι καθαρά και που εφαρμόζουν την αρχή της δέουσας υπηημέλειας. Αν η συμμετοχή είναι χαμηλή, αυτό είναι κάτι που θα ληφθεί υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν σε τρία χρόνια επανεξετάσει το θέμα και θα κάνουμε τότε κάποιες προτάσεις για να προσθέσουμε στο σύστημα κάποια υποχρεωτικά δεσμευτικά στοιχεία. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΦΚΟ. Αυτό το οποίο μας είπατε ότι το 88% των επιχειρήσεων στην παρούσα φάση δεν έχουν καμία σχέση με τους κανόνες του ΩΣΑ τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Λοιπόν, έχετε να προσθέσετε κάτι σε αυτά που είπε η προηγούμενη Γενική Διεύθυνση. Ευχαριστώ. Άλλο είναι το όνομά μου, αλλά τέλος πάντων. Ε, έχω ζήσει στις Βρυξέλλες ε, για κάποιο καιρό έχω συνηθίσει να προφέρουν το όνομά μου με όλους τους ε, δυνατούς τρόπους. Η πρόταση Νομίζω ότι πρέπει να έχετε καταλάβει ότι προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Ε, πάρα πολύ λεπτό ευαίσθητο πρόβλημα. Άρα ένας από τους πρώτους στόχους μας θα έπρεπε να είναι να μην κάνουμε την τέλεια χειρουργική επέμβαση αλλά να καταλήξει ο ασθενής. Ναι. Αυτό θα ήταν το χείριστο δυνατό σενάριο. Νομίζω ότι η λογική της πρότασης που πολύ αναλυτικά μας παρουσίασε ο συνάδελφος είναι να βρούμε την πιο σωροπημένη προσέγγιση για να πετύχουμε το στόχο μας. Χωρίς όμως υπερβολικές παράπλευρες απώλειες και παράπλευρες απώλειες θα μπορούσαν να είναι πολύ απλά το τέλος ε, του κλάδου στις αναπτυσσόμενες χώρες που όμως θέλουμε να τις υποστηρίξουμε. Επομένως υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να υιοθετήσει κανείς. Όλες αυτές τις προσεγγίσεις τις συζητήσαμε κατά την εκπόνηση της πρότασης αλλά και στο πλαίσιο του διοργανικού διαλόγου ξεκολουθούν να συζητούνται. Νομίζω όμως ότι δεν θα πρέπει να χάσουμε το βασικό στόχο και να μην ε, λησμονούμε ότι αν κάνουμε μια λάθος κίνηση εδώ μετά δεν μπορούμε να διορθώσουμε την κατάσταση. Δηλαδή όταν ε, οι προμηθευτές χάσουν κάποιους πελάτες, πολύ δύσκολα μπορούν να τους ξανακερδίσουν. Θα έχουν βρει άλλο προμηθευτή. Το δίκτυο ασφαλείας της πρότασης, όπως υπόθηκε, είναι η αξιολόγηση, αυτή η ρήτρα αξιολόγησης, όχι μετά από 10-20 χρόνια, μετά από 3 χρόνια από την έναρξη ισχύως ή τέλο από την έγκριση του κανονισμού. Άρα μπορούμε πάντοτε να αυξήσουμε τις πιέσεις. Αλλά θα είναι πιο δαπανηρό και πιο δύσκολο να επανέλθουμε εκ των υστέρων. Τα συνοδευτικά μέτρα είναι διάφορα αυτά τα μέσα, δεν χρειαζόμαστε νέα ε, μέσα και εργαλεία για τα συνοδευτικά μέτρα. Υπόκεινται στην κανονική διαδικασία προγραμματισμού αυτά τα συναδευτικά μέτρα. Στο προηγούμενο πρόγραμμα ε, ΕΤΑ ε, είχαν ζητήσει αρκετά κράτη στήριξη στον τομέα των ε, ορυχείων. Αν δεν υπάρχει ιδιοποίηση, ιδιοκτησία, αν δεν υπάρχει άνοιγμα και διαθεσιμότητα, αλλά και από την πλευρά των δικαιούχων, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σημειώσουμε πρόοδο και στα συνοδευτικά μέτρα. Βέβαια είναι δυνατόν και είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε μέτρα στον τομέα αυτό, όπως βέβαια και σε κάθε άλλο τομέα της αναπτυξιακής ε, συνεργασίας, αλλά πρέπει να έχουμε και έναν ε, συνομιλητή, έναν εταίρο. Αυτό ε, έχει να κάνει με τον πολιτικό διάλογο βέβαια. Εμείς ασκούμε μια πολύ υπεύθυνη πολιτική προγραμματισμού. Αλλά δεν μπορούμε εκ των προτέρων να ξέρουμε ποιος θα επιλέξει και ποιος θα αποφασίσει να ωφεληθεί από αυτά τα συναντευτικά μέτρα. Είναι δύο οι πλευρές που πρέπει να αποφασίσουν, είτε σε περιφερειακό είτε σε εθνικό επίπεδο. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Υπάρχει και άλλη πλευρά. Αυτά ήταν τα δύο βασικά σημεία που ήθελα να θέσω. Έγινε και μία αναφορά σε κλιμακωτούς δασμούς. Ε, δυστυχώς δεν βλέπω το βουλευτή που έκανε την ερώτηση στην αίθουσα, άρα δεν θα μακρηγορήσω. Σε ό,τι αφορά αυτή την κλιμάκωση των δασμών, ε, δεν είναι τόσο επίκαιρο αυτό, γιατί όταν μιλάμε για την Αφρική, ουσιαστικά μιλάμε για τις περισσότερες ε, από τις μη ε, ανεπτυγμένες χώρες στον κόσμο, που μπορούν αδασμολόγητα να εξάγουν όλα τα ε, εμπορεύματα, επεξεργασμένα και μη προϊόντα. Πολύ λίγη επεξεργασία, μεταποίηση γίνεται και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό, βάσιμοι λόγοι. Αλλά η κλιμάκωση των δασμών δεν είναι τόσο πρόβλημα, τουλάχιστον σε, ό,τι σε σχέση με ό,τι ίσχυε από 10-15 χρόνια. Ευχαριστώ κύριο Βένταλη, πρόεδρο. Συγητή, δεν ξέρω, θέλετε να πείτε τίποτα παραπάνω. Yes, of course. Uh, ε, βεβαίω θέλω. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Για μας το σημαντικότερο είναι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην υπολείπεται σε σχέση με τη διεθνή δηλαδή του όσα ουσιαστικά για τη δέουσα επιμέλεια. Έχει λοιπόν σημασία η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις που μου κάνατε και για τις προτάσεις σας. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Μπορώ να σας πω ότι το θέμα της πιστοποίησης Φερρυπίν και της διαδικασίας εξόριξης των μεταλλευμάτων έχει σημασία. Όχι μόνο όταν φτάνουν εδώ, αλλά όλη η αλυσίδα εφοδιασμού είναι σημαντική. Εκεί είναι το ζήτημα. Μίλησα ε, με τον εισηγητή της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, Βίνκλερ, και ελπίζω να συνεδριάσουμε οι σκιώδεις εισηγητές σύντομα για να προχωρήσουμε στην εκπόνηση της έκθεσης. Χίλια ευχαριστώ και πάλι. Σημείωσα όλες τις προτάσεις σας και προσβλέπω στην καλή μας συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Um, ευχαριστώ κύριε Βέντα, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις απαντήσεις ε, σε πολύ λεπτομερείς ερωτήσεις. Η επόμενη ανταλλαγή απόψεων θα γίνει στις 21 και 22 Ιανουαρίου με κείμενο πλέον. Θα έχουμε τη γνωμοδότηση του κύριου Βέντα ως τότε. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 29 ε, Ιανουαρίου στις 12 και η Επιτροπή μας θα ψηφίσει 24 Φεβρουαρίου και βεβαίως θα δούμε μέχρι τότε πώς θα έχει και κατάσταση των πραγμάτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή όλους σας. Θα κηρύξω τώρα τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης. Σας θυμίζω όμως ότι όταν, αν είστε συντονιστές, αύριο συνεδριάζουν οι συντονιστές στις 9. Αν δεν είστε συντονιστής θα κοιμηθείτε λίγο παραπάνω και 10.30 αρχίζει η Επιτροπή μας. Ε, με συζήτηση για την ατζέντα μετά το 2015. Η συνεδρίαση της επόμενης Δευτέρας με τον κύριο Στυλιανίδη έχει επιβεβαιωθεί για τις 5 το απόγευμα. Την άλλη Δευτέρα έχουμε βρει και αίθουσα για να ακούσουμε τον Επίτροπο κύριο Στυλιανίδη που μόλις θα έχει ε, αφιχθεί από τη Δυτική Αφρική. Παρακαλώ σημειώστε στις ατζέντες σας 5 ώρα το απόγευμα την άλλη Δευτέρα. Ευχαριστώ πολύ. Σας λέμε αύριο.